Good afternoon, everybody. Thank you for being here. Let's get started with the usual point. Καλησπέρα σε όλους. Ας ξεκινήσουμε με το σύνθεση πρώτο σημείο της σα διάταξης, δηλαδή την έγκριση της ίδιας της σα διάταξης. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρείται ως εγκεκριμένη. Το δεύτερο σημείο είναι ανακοινώσει του Προέδρου. Σε ό,τι αφορά καταρχήν τη διαρμηνία, σήμερα να πούμε ότι είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης εκτός από τα λετωνικά και τα αγγέλικα ελληνικά. Επίσης υπάρχει βέβαια για το σύνθεση σημείο της έγκρισης των συμπερασμάτων των συντονιστών και έχουμε και τον διορισμό των εισηγητών. Καταρχήν, μία πρόταση σε ό,τι αφορά έκθεση σε σχέση με τον σοβαρό κίνδυνο τη ε, παραβίαση του κράτου δικαίου από την πλευρά τη Πολωνία, ε, το οποίο έχω αναλάβει εγώ. Μετά, δεύτερο, διορισμό εισηγητών σε ό,τι αφορά γνωμοδότηση. Και συγκεκριμένα η κυρία Τέρι Ρέγκε έχει διοριστεί ω εισηγητή για την γνωμοδότηση τη ΛΥΜΠΕΣ σε ό,τι αφορά τι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο, σε ό,τι αφορά ε, την εμηνία του προπολογισμού σε περίπτωση που υπάρχουν ε, λήψεις και την τήρηση του κράτους δικαίου. Αυτοί λοιπόν είναι διορισμοί ε, που προτείνονται σε ό,τι αφορά τους εισηγητές. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα λοιπόν με, αυτές, με αυτούς τους διορισμούς και αυτές τις ανακοινώσεις θεωρούμε πως εγκρίνονται. Και μετά το σημείο 3 της, των ανακοινώσεων εδώ είναι η κατεξοδότηση. εκτελεστικές πράξεις, όσες εκτελεστικές λοιπόν πράξεις έχουμε μια εκτελεστική απόφαση, τροποποίηση, μια άλλη τροποποιητική απόφαση σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα εργασία, εργασιών του 2018 και τη χρηματοδότηση δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, αρρωγής έκτακτης ανάγκης σε ό,τι αφορά το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Ε, και εδώ έχουμε να κάνουμε με το γεγονός ότι ε, η εφαρμογή αυτής της εκτελεστικής πράξης κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη της ΛΥΜΠΗ μέσω του ενημερωτικού δελτίου του newsletter, δηλαδή της ΛΥΜΠΗ. στις 11 Οκτωβρίου και η προθεσμία για την εκφράση οποιοδήποτε αντιρρήσεων έχει οριστεί ως 22 Οκτωβρίου. Και μετά υπάρχει σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της ε, Επιτροπής σε ό,τι αφορά το ε, πρόγραμμα χρηματοδότησης και το πρόγραμμα εργασιών του 2020 και η λήψη αυτής της εκτελεστική πράξη ανακοινώθηκε και πάλι σε όλα τα μέρη τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ μέσω του ενημερωτικού δελτίου τη Επιτροπή τη 11 Οκτωβρίου. Και η εσωτερική προθεσμία για την έκφραση αντιρρήσεων έχει οριστεί και πάλι ως 22 Οκτωβρίου. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τις ανακοινώσεις του Προέδρου. Και περνάμε τώρα στα ουσιαστικά σημεία της σημερινής διάταξης και συγκεκριμένα τα ζητήματα που θα συζητήσουμε σήμερα. Ξεκινάμε λοιπόν με το σημείο 3 της σημερινής διαταξή, που είναι ο Frontex, Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Η κυρία Μετσόλα είναι εδώ, συγγήτριά μα. Ε, και εδώ ουσιαστικά θα εξετάσουμε μόνο και μόνο ένα διορθωτικό, τίποτα άλλο. Έχουμε να κάνουμε εδώ με μια σημαντική νομική πράξη για την οποία όλες οι πολιτικές διεργασίες έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της προηγούμενης θητείας του, του Κοινοβουλίου, 2014-2019. Και στο πλαίσιο των συζητήσεων και των συμπερασμάτων που, ή μάλλον ε, δεν ήταν δυνατό ωστόσο να ολοκληρωθούν οι συζητήσει και να αντιληφθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα στο πλαίσιο τη προηγούμενη θητεία σε ό,τι αφορά το πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, ε, που προβλέπει μεταξύ άλλων και ένα μόνιμο σώμα 10.000 συνοριοφυλάκων. Και αυτό είναι και το βασικό ζήτημα σε ό,τι αφορά την ε, αναθεώρηση ε, του ε, κανονισμού για τον Frontex. Η αναθεώρηση λοιπόν από τους νομοσωμαθείς νομικούς δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της προηγούμενης ε, κοινοβουλευτικής εθιτείας και γι' αυτό λοιπόν υποβλήθηκε τώρα, υποβλήθηκαν αυτές οι τροποποιήσεις με τη μορφή διορθωτικού και ανακοινώθηκε σε όλα τα μέλη ε, της ΛΥΜΠΕ και σε όλες τις γλώσσες την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε να κάνουμε απλώς και μόνο με ένα τεχνικής φύσης διαδικαστικό ζήτημα σε σχέση με αυτό το ζήτημα το οποίο μας αφορά και θα δώσω το λόγο στην συγγήτρια την κυρία Μετσόλα για να μας παρουσιάσει το λόγο διορθωτικό. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μία αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής ε, Ακτοφυλακής και Συνοριοφυλακής πέρυσι. Μέσα σε έξι μήνες καταφέραμε να φτάσουμε, να κάνουμε το αδύνατο. Συμφωνήσαμε μεταξύ μας. Υπήρξε πλειοψηφία εντός των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταφέραμε να συμφωνήσουμε επίσης επί Ρουμανικής Προεδρίας και τώρα επί Φιλανδικής Προεδρίας. Καταφέραμε να συμφωνήσουμε επί του φακέλου και να τον υπερψηφίσουμε λίγο πριν ολοκληρωθεί η προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Με βάση τη διαδικασία θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το φάκελο αυτό, ούτω ώστε να μην υπάρχουν λάθη. Αυτό τι σημαίνει. Ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις Έγιναν μάλλον κάποιες διευκρινήσεις και αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξουμε την αρρύθμιση κάποιων παραγράφων λόγω του ότι υπήρξαν κάποιες ε, διορθώσεις και κάποιες απαλληφές στο κείμενο. Αυτή η διαδικασία δεν μπορούσε να γίνει πριν την ε, ψηφοφορία στην Επιτροπή Λίμπε και στην Ολομέλεια, γιατί απαιτεί πάρα πολύ χρόνο. Αυτή η αναθεώρηση δηλαδή ήταν πολύ χρονοβόρα και γι' αυτό μπορέσαμε να σας παρουσιάσουμε αυτό το φάκελο, το διορθωτικό δηλαδή φάκελο, μόλις σήμερα ε, πάνω στο θέμα της ε, Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής και Συνοριοφυλακής. Με αυτή λοιπόν την παρουσίαση του διορθωτικού ολοκληρώνουμε την νομοθετική διαδικασία και ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ τις επόμενες εβδομάδες. Ούτω ώστε ο οργανισμός να αρχίζει να εφαρμόζει αυτό τον κανονισμό. Ήταν πολύ σημαντικό να συμφωνήσουμε τον περασμένο Μάρτιο από πολιτική άποψη και καταλήξαμε ότι ο οργανισμός, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ακτοφυλακής και Συνοριοφυλακής θα έχει 10.000 συνοριοφύλακες ούτω ώστε να διεκπεραιώνει το πολύ εκτενές και σημαντικό έργο του. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Frontex έχει ενισχυθεί και έχουμε εισαγάγει και ασφαλιστικές δικλείδες ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Έχουμε δώσει μεγαλύτερη σημασία στα θεμελιώδη δικαιώματα και έχουμε βελτιώσει τον μηχανισμό υποβολής ε, παραπόμνων και υπάρχουν τώρα και οι παρατηρητές ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιωδών δικαιωμάτων που θα παρακολουθούν τις δραστηριότητες της Frontex για να δούμε, είμαστε σίγουροι ότι τηρούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτή η γλωσσική αναθεώρηση του κειμένου δεν έχει αλλάξει ουδόλω στην ε, πολιτική συμφωνία στην οποία είχαμε φτάσει. και σε ό,τι συμφώνησαν οι ευρωβουλευτέ στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Τίποτα από αυτά δεν έχει αλλάξει. Η αλλαγή αφορά το άρθρο 73 που μιλούσε, αναφερόταν μάλλον σε μία παράγραφο που δεν υπήρχε. Διορθώθηκε αυτό το λάθος. Επίσης, στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 72 έχουμε εισαγάγει μια νέα διατύπωση που ξεπερνούν τις διμερείς ε, συμφωνίες. Αυτό το σημείο δεν υπήρχε πριν σε αυτό το άρθρο. Υπήρχαν και άλλες παραλήψεις επίσης και έχουν διορθωθεί όλα αυτά. Επίσης, σε διάφορα άρθρα είχαμε παρατηρήσει ότι αναφερόμαστε σε κάποιες έννοιες όπως τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων ή τον έλεγχο των συνόρων. Ή σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούσαμε το should αντί για το shall, το θα πρέπει αντί για το πρέπει. Άλλους χρόνους, λάθος χρόνους. Επίσης, διορθώσαμε τη φρασιολογία και οποιαδήποτε αναφορά κάναμε στο προσωπικό, ούτω ώστε να χρησιμοποιούμε τη σωστή ορολογία παντού. Αυτό το έγγραφο έχει αλλάξει ως προς κάποια τεχνικά σημεία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αλλάζει την πολιτική συμφωνία στην οποία είχαμε φτάσει. Το σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε ότι η εφαρμογή αυτού του κανονισμού γίνεται απρόσκοπτα και ότι η πολιτική συμφωνία που έφτασε το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Κομισιόν και το Συμβούλιο αρχίζει να ισχύει, ούτω ώστε να ενισχύσουμε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ την κυρία Μετσόλα για την ενδελεχή εξέταση, ε, εξήγηση της όλης κατάστασης. Είναι τεχνικό το θέμα. Υπήρχαν κάποια τεχνικά ζητήματα που διορθώσαμε. Σα δόθηκαν τεχνικές εξηγήσει, ορίστε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σχόλια. Να τα ακούσουμε. Εάν όχι... Yes, we, may accept the, the, the Μπορούμε λοιπόν να αποδεχθούμε το διορθωτικό αυτό παράρτημα. Ο κανονισμός μας δίνει τη δυνατότητα να το κάνουμε, είναι απολύτως θεμητό και νόμιμο είναι μια διόρθωση Συνεπώς αποδεχόμεστα λοιπόν τις εξηγήσεις σας. Εξετάσαμε την προσθήκη, τη διορθωτική αυτή προσθήκη κατανοήσαμε το λάθος το οποίο επισυνέβη και το οποίο ε, θα πρέπει να διορθωθεί με τον ορθό τρόπο όπως ακριβώς προβλέπεται από τον κανονισμό μας. Γι' αυτό λοιπόν και η υπηρεσία λειτουργίας της Ολομέλειας θα ανακοινώσει στην επόμενη μήνυ Ολομέλεια των Βρυξελών ε, ή όχι στο Στρασβούργο τελικά θα ανακοινώσει τη διόρθωση αυτή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για το συγκεκριμένο σημείο, τελειώσαμε με αυτό. Είδαμε ότι το επόμενο θέμα, θέματα ε, εσωτερικών υποθέσεων και δικαιοσύνης, ανταλλαγή απόψεων ε, με την Επιτροπή και το Συμβούλιο σε 10 λεπτά. Γι' αυτό λοιπόν υπολογίσαμε περισσότερο χρόνο από ό,τι είχαμε ανάγκη και γι' αυτό λοιπόν για να μπορέσουμε να δώσουμε την δυνατότητα να είναι παρούσα η Επιτροπή και το Συμβούλιο διακόπτουμε για 10 λεπτά παρακαλώ εφόσον συμφωνείτε. for Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν. Θα μας παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν τα θέματα τα εσωτερικά. Την προηγούμενη εβδομάδα οι Υπουργοί Δικαιοσύνη συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο αρχές Οκτωβρίου για να συζητήσουν τα θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως και στο παρελθόν, το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν ανταλλάξει απόψεις στα θέματα αυτά ιδιαίτερα σε ορισμένες περιπτώσεις όπου τα θέματα αποκτούν υψηλή θα έλεγα επικαιρότητα και προτεραιότητα. Καλωσορίζω λοιπόν την Προεδρία του Συμβουλίου και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να μας εκθέσουν τα θέματα τα οποία συνεζήτησαν στην τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων από την Προεδρία του Συμβουλίου. Έχουμε την κυρία Βάκουρη από το Υπουργείο Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Φιλανδίας και την κυρία Κατήλα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε τον Γενικό Διευθυντή κυρία Παρασκευή Μίχου, εσωτερικές υποθέσεις, όπως επίσης και την κυρία Στόλα από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης. Θα ήθελα τώρα να κάνω μία μικρή εισαγωγή, αν θέλετε. Έχουμε να κάνουμε με πάρα πολλά θέματα. Νομίζω ότι το Συμβούλιο θα αναφερθεί στα θέματα στα εσωτερικά, στην έρευνα και αναζήτηση, και την χρήση των νέων ε, τεχνολογιών για, τα, για τη δικαιοσύνη, κοινέ αξίες, ανθρώπινα δικαιώματα, θεμελιώδη δικαιώματα και δράσεις εναντίον της διαφθοράς. And answers to our guest Νομίζω ότι όλα αυτά θα μας βοηθήσουν να αποκτήσουμε μια καλύτερη εικόνα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το Συμβούλιο, με την Προεδρία, από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης παρακαλώ και μετά θα ακολουθήσουμε και την Γενική ε, Διεύθυνση Δικαιοσύνης. Δεν έχει έρθει ακόμα η κυρία Μίχου. Θα της δώσουμε λοιπόν λίγο χρόνο και θα ξεκινήσουμε με τα θέματα της δικαιοσύνης μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η κυρία Καρτίλα έχει το λόγο για 12 λεπτά και ήρθε η εκπρόσωπος, η Γενική Διευθύντρια. Αγαπητά μέλη, σας ευχαριστώ που μου προσκαλέσατε σήμερα να σας παρουσιάσω τις συνεχιζόμενες εργασίες του Συμβουλίου στον τομέα της δικαιοσύνης, τον Φιλανδικό. Ο Η Φιλανδή υπουργό, η κυρία Χέντριξεν, εξέθεσε τις προτεραιότητες ε, τον Σεπτέμβριο της ε, Προεδρίας μας και εξέθεσε επίσης και τις υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνουμε γύρω από το θέμα του σεβασμού των ευρωπαϊκών αξιών. Το κράτος δικαίου είναι ε, το σημείο στο οποίο εδράζεται η συνεργασία των κρατών μελών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει συνεισφέρει τα μάλα στην πορεία της μέχρι τώρα. Το θέμα αυτό παραμένει βασική προτεραιότητα και για μας τους Φίλανδους. Προσπαθούμε να βρούμε πιο αποτελεσματικούς τρόπους έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες στα κράτη-μέλη και να υπογραμμίσουμε τα, τα πιθανά προβλήματα και να βρούμε τρόπους καταπολέμησης επίσης της διαφθοράς μέσω του σεβασμού των αξιών και της αύξησης της εμπιστοσύνης των πολιτών στις δημόσιες αρχές. Υπουργοί Δικαιοσύνης <clears throat> τα συζήτησαν τα θέματα αυτά εδώ και μία εβδομάδα και υπάρχουν τρεις τομείς που θα μου επιτρέψετε να σημειώσω σαν βήματα προόδου. Πρώτον, το Συμβούλιο επιβεβαίωσε την υποχρέωση την οποία έχει για να συνεχιστεί η διαδικασία συμμετοχής πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της στην ε, ε, Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Θεωρούμε ότι είναι ένας ελίπων κρίκος για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ένωση. Ε, οι προσπάθειες έχουν ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια και εμείς απλά συνεχίζουμε την διαδικασία αυτή και ελπίζω να ολοκληρωθούν με επιτυχία στο μέλλον οι προσπάθειες. Ε, επίσης θα κάνουμε ορισμένες προτάσεις και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πιθανές οδηγίες σε τα επόμενους μήνες. Δεύτερον, τώρα για την χάρτα των, ανθρωπίνων δικαι... των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ένα νομικά δεσμευτικό όργανο εδώ και 10 χρόνια είναι αναπόσπαστο τμήμα της ε, θεσμικής αρχιτεκτονικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να γίνεται σεβαστό. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν προκλήσεις στον τομέα της έλλειψης και καταπολέμησης των διακρίσεων και το Συμβούλιο θα συνεχίσει την προσπάθεια καταπολέμησης κάθε μορφής διάκρισης. Η κοινωνία των πολιτών και οι εκπρόσωποι της έχουν ένα σημαντικό ρόλο να παίξουν εδώ για τις μελλοντικές εργασίες μας στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, το Συμβούλιο αναλαμβάνει την υποχρέωση ετησίου διαλόγου και ανταλλαγής χρηστών πρακτικών σε εθνικό επίπεδο. Οι Υπουργοί έχουν συζητήσει επίσης και τις μελλοντικές προκλήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα ένα από τα θέματα που συζητήθηκε ήταν η διάδοση των θεμελιωδών αρχών. Πολλές φορές θεωρούνται δεδομένες οι αρχές αυτές. Ε, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων ετέθησαν θέματα, το θέμα της ψηφιοποίησης και της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο. Και τέλος, στην τελευταία συνάντηση της Δευτέρας, στρέψαμε την προσοχή μας στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Συζητήσαμε πολλαπλές μορφές α, της διαφθοράς στα πλαίσια των προτάσεων της Προεδρίας. Η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι αναπόσπαστο τμήμα μιας ευρύτερης προσπάθειας που ξεκίνησε τον Ιούλιο στο Ελσίνκι το Ιούλιο είχαμε μια συζήτηση και για τον ρόλο των Υπουργών Δικαιοσύνης στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στον σεβασμό του κράτους δικαίου. Είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί στο σύνολό του σε κάθε κράτος μέλος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την αμοιβαία πλήρη εμπιστοσύνη μεταξύ μας η μεγάλη πλειοψηφία των υπουργών συμφωνούν να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική. Πολλοί υπουργοί υπογράμμισαν την ανάγκη που υπάρχει για την Ευρώπη να προσθέσει αξία εδώ, να δημιουργήσει προτιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Χρειάζεται περισσότερη μορφή συνέργειας και επικοινωνίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ε, να ανήκει το θέμα της καταπολέμησης της διαφοράς στο σύνολο των συζητήσεων για το κράτος δικαίου. Θα πρέπει να λειτουργήσουμε υποδειγματικά σε, ε, στη διεθνή σκηνή. E έχουμε συνδέσει, συνδεθεί έτσι και αλλιώς ε, με τη σύμβαση Γκρέκο και θα έχουμε αναλάβει την υποχρέωση να γίνουμε σε κάποια φάση επόμενη πλήρη μέλη. Ε, νομίζω ότι εδώ συνεργαζόμαστε και με τις προσπάθειες τις οποίες κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και ένα τελευταίο σημείο θα ήθελα να υπενθυμίσω αυτά τα οποία η Υπουργό Δικαιοσύνης της Φιλανδίας σας είπε τον μήνα Σεπτέμβριο. Παρατήρησε ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα τύχουν ε, ειδική προσοχής, όπως η διαφάνεια. Πολλά θέματα την προηγούμενη εβδομάδα είχαν ε, αυτό το αντικείμενο, καταπολέμηση, θεμελιώδη δικαιώματα, διαφάνεια. Πιστεύουμε ότι ε, διαδικασίες λήψεως αποφάσεων διαφανέστερες θα φέρουν τους πολίτες πολύ πιο κοντά ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για τη συνεργασία σας και ελπίζουμε να συνεχιστεί. Ευχαριστώ την εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, η κυρία Στόλα. Ε, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση για να συζητήσουμε στην ΛΥΜΠΕ τα αποτελέσματα του τελευταίου Συμβουλίου Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων. Χαίρομαι πάρα πολύ που έρχομαι για πρώτη φορά ενώπιον τη ΛΥΜΠΕ ε, στην έκνο βουλευτική θητεία. Ε, Γενική Διευθύντρια είμαι για θέματα δικαιοσύνη και ως, ε, υπό αυτή την ιδιότητα θέλω να σα εκφράσω την απόλυτη διάθεσή μου να συνεργαστούμε για τα θέματα τη αρμοδιότητά μα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τους Ευρωπαίους πολίτες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και την Προεδρία για την ε, πολύ εποφελή συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών περασμένη εβδομάδα. Καταρχά, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρθηκε ήδη από την κυρία Μάρια Κάρτιλα. Καλωσορίζω τη συμφωνία για το όνομα του πρώτου Ευρωπαίου Εισαγγελέα, του Άρχη Εισαγγελέα και θέλουμε να διοριστεί το συντομότερο δυνατόν. Ε, υπάρχει πρόοδος στη δημιουργία και σύσταση του γραφείου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα θα πρέπει η αρχή εισαγγελέα να αναλάβει τα καθήκοντά τη, αλλά και το σώμα των εισαγγελέων να αρχίσει να λειτουργεί. Γι' αυτό η Κομισιόν καλεί τα κράτη-μέλη που δεν έχουν προτείνει υποψηφίου ε, για το αξίωμα του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα να το κάνουν το συντομότερο δυνατό. Ένα άλλο σημαντικό είναι τα κράτη-μέλη να κάνουν τι απαραίτητε προσαρμογέ στα, ε, στην εσωτερική θάση και να εφαρμόσουν την οδηγία για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη λεγόμενη PIF. Έχουμε στείλει προειδοποιητικά γράμματα και επιστολές στα κράτη-μέλη, τα οποία δεν έχουν κοινοποίησει την ενσωμάτωση στην εσωτερική τάξη της νομοθεσίας του νομοθετήματος PIF και συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη για να τα βοηθήσουμε να την εφαρμόσουν. Το Συμβούλιο υιοθέτησε συμπεράσματα για το Eurojust, τα οποία υποστηρίζουμε πλήρως. Όπως ξέρετε, ο νέος κανονισμός για το Eurojust θα εφαρμοστεί από τις 12 Δεκεμβρίου του 19 και το νέο νομικό πλαίσιο θα επιτρέψει στο Eurojust να αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά ε, τους φακέλους για θέματα εγκλήματος όπως ε, τρομοκρατία, σωματεμπορία, διακίνηση ανθρώπων, ε, διακίνηση μεταναστών, κυβερνοέγκλημα, διαφθορά. Υπάρχει ένα μητρό για την ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Υπάρχει ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε τις τελευταίες ψηφιακέ τεχνολογίε για την δικαστική συνεργασία και η Κομισιόν ξεκίνησε μία έρευνα για να δούμε τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε στον τομέα αυτό. Στην Συνεδρίαση του Συμβουλίου ενημερωθήκαμε για τι πρώτε επίσημε διαπραγματεύσει ε, με τις ΗΠΑ για τα, την ηλεκτρονική λήψη ε, αποδεικτικών στοιχείων. Έγινε ο πρώτο γύρο. Ε, θα σα ενημερώνουμε τακτικά σε όλε τι φάσει των διαπραγματεύσεων για το πώ προχωρούν αυτέ. Αυτή η πρώτη συνάντηση ήταν μια ευκαιρία για κάθε πλευρά για να εξηγήσει ποια είναι το σημείο αφετηρίας της. Η Κομισιόν ξεκαθάρισε ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις γίνονται με βάση μια δημόσια εντολή που έχει δώσει το Συμβούλιο για την πρόταση για τη λήψη ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων. Η Κομισιόν ξεκαθάρισε ότι η θέση της στις διαπραγματεύσεις εξαρτάται από το πώς εξελίσσεται το πακέτο για την, ε, τα, τις εσωτερικές υποθέσεις, νομοθετικός πώς. Η κυρία Σίπελ είναι η εισηγήτρια του Κοινοβουλίου και την καλούμε να ξεκινήσει την κοινοβουλευτική διαδικασία των συντομότερων δυνατών. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι έχει μια εντολή για να διαπραγματευτεί την ε, ευρωπαϊκή ε, συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων αφορούσε πολλά βασικά θέματα, τα είδη των ε, δεδομένων, ε, κυρώσεις, αρμόδιες αρχές, άχθος εργασίας και ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία δεδομένων. Συμφωνήσαμε με τους ε, Αμερικανούς ομολόγους μας να αναπτύξουμε περαιτέρω ε, και να διερευνήσουμε περαιτέρω σε συζητήσει στα θέματα αυτά. Ένα δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων πρόκειται να γίνει στι 6 Νοεμβρίου και ο στόχο είναι να σημειωθεί συγκεκριμένη πρόοδο πριν από την Υπουργική Ευρωπαϊκή Ένωση είπα, το Δεκέμβριο. Η Μαρία Κάρτιλα ανέφερε τα θέματα που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και την πρόσβαση στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, την προσχώρηση μάλλον στο Συμβουλίο της Ευρώπης, καθώς και τις συμπληρωματικές οδηγίες για αυτά τα θέματα, καθώς και τη χάρτα. Θα ήθελα να αναφέρω επίσης τη συζήτηση που έγινε για την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας για την καταπολέμηση ρητορίας μίσους ε, στο διαδίκτυο. Και να σας δώσω κάποιες πληροφορίες, γιατί νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που συζητάμε αυτό το θέμα στη ΛΥΜΠΕ. Αυτός ο κώδικας δικαι... ε, δεοντολογίας ε, υπογράφηκε το Μάιο του 2016 και καλύπτει 96 από τις ε, πλατφόρμες ε, online που υπάρχουν που μπορούν να επηρεάζονται από τέτοιες ρητορικές. Αυτός ο κώδικας διοντολογίας βασίζεται σε δύο διαφορετικούς πυλώνες. Ο πρώτος είναι η προειδοποίηση και δράση. Όταν μία προειδοποίηση για παράνομο λόγω μίσους ε, λαμβάνεται, τότε η εταιρεία θα πρέπει να εξετάζει ε, το συγκεκριμένο αυτό σημείο εντός 24 ωρών και να το διαγράφει. Και υπάρχει και ένας μηχανισμός ε, συνεργασίας μεταξύ των εταιριών, των εθνικών αρχών, των οργανώσεων το, της κοινωνίας των πολιτών, δεύτερος πυλώνας, για να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές προκλήσεις της ρητορικής μίσους και να βοηθήσουμε τις διοκτικές αρχές. Υπάρχει πρόοδο. Το 2016 μόνο το 28% του περιεχομένου αυτού αφαιρούνταν και τώρα έχουμε φτάσει στο 72%. Επιπλέον, 89% των προειδοποίησεων εξετάζονται εντός 24 ωρών, ενώ προηγουμένως ήμασταν πριν τον κώδικα, δηλαδή στις 40, στις 40 ώρες. Επίσης, ε, οι πλατφόρμες έχουν περισσότερο προσωπικό που εξετάζει αυτό το περιεχόμενο και απαντάει στις προειδοποίησεις, καθώς και πληροφορίες για το κοινό ε, όταν λαμβάνονται δράσεις εναντίον των ρητορικών μίσους. Σε σχέση με τη συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι εταιρείε IT από το 2016 έχουν δημιουργήσει ένα δίκτυο ε, με νοικιό εμπιστοσύνη για να προωθήσουν ε, αφηγήματα κατά τη ρητορία μίσου. Ο κώδικα ε, αυτό δημιούργησε ένα περιβάλλον αμοιβαία ε, εμπιστοσύνη, ανταλλαγή γνώση και συνεργασία και γι' αυτό έχουμε αυτά τα γρήγορα αποτελέσματα. Όμω, θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την πρόοδο και να παρακολουθούμε του σύνεγγυ στην κατάσταση στο μέλλον, λαμβάνοντα υπόψη τι εθνικέ επίση πρωτοβουλίε. Οι νέε προκλήσει, όπω η σχέση που έχουν οι εξεμιστικές ομάδες με αυτούς που γράφουν αυτές τις ρητορικέ. Ε, καθώς με ακροδεξιούς, ε, ε όλες αυτές οι σχέσεις θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω. Ο κώδικας διοντολογίας είναι μια πρωτοβουλία αυτορύθμισης που συμπληρώνει τη δουλειά που θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο εφαρμογής ε, νόμου που καταπολεμούν την ξενοφοβία και το ρατσισμό. Έχουμε ενημερώσει επίσης με την ανακοίνωση για το EGDPR ε, για θέματα ΛΟΑΔ με βάση ε, τη συζήτηση που έγινε στις Βρυξέλλες 23 και 24 του μηνός. Ναι, και τώρα θα ακούσουμε και την άποψη από την πλευρά της Γενικής Διεύθυνσης HOME και την αντιπροσωπεία εδώ του ε, Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τα ζητήματα εσωτερικών υποθέσεων είναι η, ε, τα όσα θα ακούσουμε τώρα για να ολοκληρώσουμε την άποψή μας ε, για να ακούσουμε και ποια ήταν τα τελευταία συμπεράσματα του Συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων. Θα ακούσουμε λοιπόν την Ειρή Βακούρη καταρχήν για, την, για το Συμβούλιο και μετά την κυρία Μισού από την Γενική Διεύθυνση Την κυρία Μίχου, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστούμε που προσκαλέσατε τη Φιλανδική Προεδρία στη σημερινή σα συνεδρίαση ε, για να αναφερθούμε ακριβώς στα ζητήματα των ιστορικών υποθέσεων. Όπως ε, είναι γνωστό και όπως αναφέρθηκε και από την ε, Υπουργό κυρία Μαρίσαλο που ήταν μπροστά και βρέθηκε εδώ ενώπιον τη συνεδρίασής σα. Αυτή τη στιγμή έχουμε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς ολοκληρώνεται ο θεσμικός κύκλος και κατά συνέπεια θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να κάνουμε ένα προβληματισμό και να ε, συζητήσουμε το μέλλον του τομέα των εσωτερικών υποθέσεων εις βάθος. Και αυτό μας το επιτρέπουν και ε, νομοθετικοί φάκελοι του οποίου εξετάζουμε αυτή την ε, περίοδο. Θα ήθελα τώρα να εστιάσω σε, τρεις, σε τρία ζητήματα τα οποία θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικά και επίκαιρα από την πλευρά τη Φιλανδική ε, Προεδρία στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων. Θα ξεκινήσω από τη μετανάστευση και τι επιχειρήσει έρευνα και διάσωση που ήδη αναφέρθηκαν από τον Πρόεδρο. Οι εξελίξει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και στι αρχέ του φθινοπόρου ανέδειξαν μία σειρά από ανησυχίε σε ό,τι αφορά τις ε, τρεις κύριες μεταναστευτικές οδούς για τις Μεσογείου. Καταρχήν παρατηρούμε αύξηση των ε, αφήξεων στα ελληνικά νησιά. Το Σεπτέμβριο δηλαδή ε, τις 11.500 αφήξεις στην Ελλάδα. Δηλαδή από τότε που άρχισε να εφαρμόζεται η δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, Τουρκία είναι ο ψηλότερος μηνιαίος αριθμός ε, και η Ελλάδα έχει ήδη λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσει αυτέ τι αυξημένε προκλήσει μεταξύ αυτών και σχέδια για την αναθεώρηση των, της νομοθεσίας ασύλου αλλά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στα hot spots. Επίση, υπάρχουν και κάποια μέτρα προκειμένου να αυξηθούν οι επιστροφέ. Τώρα, η Επιτροπή και οι υπηρεσίε τη εξετάζουν τρόπου για να παράσχουν περισσότερη υποστήριξη. Και βρισκόμαστε σε κατάλληλη χρονική συγκυρία για να δούμε πώ τα κράτη-μέλη μπορούν από την πλευρά του να ε, παράσχουν περισσότερη υποστήριξη. Πέραν τώρα τη Ελλάδα, θα πρέπει να εξετάσουμε και τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο. καθώς έχουμε περισσότερες αφήξει από την Τουρκία θα επανεξετάσουμε και την ε, παροχή αρρωγή που προσφέρουμε στην ε, Τουρκία. Όλοι μας ε, γνωρίζουμε πως κατά τελευταία χρόνια η Τουρκία έχει δεχτεί υψηλέ μεταναστευτικέ πιέσεις και στα δικά τη σύνορα. Και τα πράγματα τώρα, όπως μαθαίνουμε όλοι μας από τις ειδήσει, έχουν εξελιχθεί περαιτέρω. Υπάρχει μια περαιτέρω δηλαδή καμπή εδώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο συγκεκριμένα θα εξετάσει εν λόγω ζήτημα αυτή την εβδομάδα. Όπως γνωρίζετε υπάρχει μια ε, συμφωνία μεταξύ τεσσάρων κρατών μελών της Ιταλίας, της Μάλτας, της ε, Γερμανίας και της Γαλλίας ε, σε ό,τι αφορά τις αφήξει στην κεντρική Μεσόγειο. Κατά την άποψη της Φινλανδίας αυτή η συμφωνία αποτελεί ουσιαστικά ένα πρώτο βήμα στο να έχουμε πιο προβλέψιμες αφήξεις από τη θάλασσα, στο πλαίσιο δηλαδή και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Καθώς αυτή η συμφωνία βέβαια είναι περιορισμένη σε ό,τι αφορά τη χρονική της διάρκεια και έχει περισσότερο πιλωτικό χαρακτήρα, παρόλα αυτά παραμένει σημαντικά και από πρακτική αλλά και από ανθρωπιστική άποψη. Δηλαδή πολλοί από τους ανθρώπους οι οποίοι διασώζονται ε, στη Μεσόγειο έχουν κακή κατάσταση υγείας και οι διαδικασίες λοιπόν για την άφηξή τους ε, διασφαλίζουν τη μη περαιτέρω επιδείνωση της υγείας τους. Ε, και βέβαια θα πρέπει σιγά σιγά να ε, ξεφύγουμε από την προσέγγιση της μετεπιβίβασής τους από πλοίο σε πλοίο και να κινηθούμε σε πιο προβλέψιμες εγκαταστάσεις. Και θα πρέπει βέβαια να έχουμε ένα πιο οργανωμένο πλαίσιο και όχι ad hoc ε, επιμέρους δηλαδή λύσεις. Ε, και η Φιλανδική Προεδρία έχει προτίμησει όλα τα κράτη-μέλη να εξετάσουν την δυνατότητα συμμετοχή τους ε, σε αυτή τη συμφωνία. Με ένα μεγαλύτερο δηλαδή αριθμό κρατών που θα συμμετείχαν, το εν λόγω πιλωτικό project θα μπορούσε να είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο σε ό,τι αφορά και την υποβοήθηση των, των χωρών γενικά που δέχονται αυτές τις πιέσεις και προκειμένου να έχουμε περισσότερες βάσεις για τη μελλοντική αναθεώρηση του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι όταν και εφόσον επιτύχουμε κάποια πρόοδο σε κάποια από αυτέ τι μεταναστευτικέ οδού, παρόλα αυτά αυτό δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε τι εργασίε που κάνουμε σε ό,τι αφορά τι υπόλοιπε οδού. Δηλαδή, προτεραιότητα για μα παραμένει τα κράτη εκείνα τα οποία βρίσκονται υπό σε όλη την Ευρώπη να λαμβάνουν υποστήριξη μέσω κοινών προσπαθειών. Τώρα, υπάρχουν δύο ακόμα σημεία στα οποία θα ήθελα να αναφερθώ σήμερα είναι κατα... κυβερνοαπειλές και στη συνέχεια οι νέες τεχνολογίες. Τώρα, η υψηλότερη ετοιμότητα σε ό,τι αφορά... Η, και τα όσα αναφέρονται και στην ε, ατζέντα μας καταδεικνύουν το πόσο, το πόσο σημαντικό είναι να ε, έχουμε περισσότερη ετοιμότητα σε ό,τι αφορά αυτές τις ε, τις κυβερνοαπειλέ. Χρειαζόμαστε περισσότερου πόρου και περισσότερε τεχνολογικέ ικανότητε για να το επιτύχουμε αυτό. Όλε οι συζητήσει που κάναμε μέχρι τώρα στα διάφορα προπαρασκευαστικά σώματα του Συμβουλίου και σε υπουργικό επίπεδο έχουν καταδείξει ότι υπάρχουν περιθώρια και υπάρχει ανάγκη για την υιοθέτηση μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για την υποστήριξη των κρατών μελών προκειμένου να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδου απειλέ. Ε, για την αντιμετώπιση αυτού του είδου απειλών σε επίπεδο εσωτερική ε, πολιτική. Βέβαια, κυρίω αρμόδια είναι τα κράτη-μέλη, αλλά παρόλα αυτά χρειάζονται συμπληρωματικέ ευρωπαϊκέ δράσει. Η ε, σημασία λοιπόν ε, μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την μετώπιση τέτοιων απειλών είναι, είναι κάτι το οποίο έχει αναγνωριστεί και για παράδειγμα διαρροή κάποιων ε, ψευδών ε, βίντεο μπορεί να έχει ε, πολύ σημαντικές ε, επιπτώσεις. Δημιουργούν δηλαδή προβλήματα σε ό,τι αφορά τις εργασίες και των αστυνομικών αλλά και άλλων αρχών προστασίας και μπορούν να υπάρξουν δηλαδή συναισθήματα σε ό,τι, όπως θυμός, όπως πανικός και άλλα και δεν επιτρέπουν την ψύχρεμη αντιμετώπιση ε, των καταστάσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τρίτο σημείο και τι νέε τεχνολογίε, θα πρέπει εδώ να παρακολουθούμε, στο πλαίσιο δηλαδή τη εσωτερική πολιτική τη Ένωση, το τι συμβαίνει σε σχέση με τι νέε τεχνολογίε. Η Φιλανδική Προεδρία ε, δίνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το ζήτημα και ο γενικότερο στόχο μα είναι να αναλάβουμε έναν ενεργό ρόλο εδώ αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που μας παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, αλλά προβλέποντας ταυτόχρονα και περιορίζοντας τους δυνητικούς κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Οι νέε αυτέ τεχνολογίε επηρεάζουν όλε τι αρχέ και όλε τι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι συναρμόδιε για την προστασία τη ε, ασφαλεία μα. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι αρχέ μα και οι επιχειρησιακέ του αρχέ λαμβάνονται υπόψη όταν ε, αναπτύσσουμε νέες τεχνολογίες όπως ε, το 5G. Ε, γιατί θα υπάρξουν μία σειρά από επιπτώσεις σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την ασφάλεια των δεδομένων αλλά και τις κρίσιμες υποδομές. Η κοινή αξιολόγηση κινδύνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 5G και η νέα εργαλειοθήκη, το Toolbox, θα παίξουν εδώ ένα σημαντικό ρόλο για την εξασφάλιση τη απαραίτητη προστασία των δικτύων μα. Η Φιλανδική Προεδρία θεωρεί πω είναι σημαντικό να οθετήσουμε μια συντονισμένη προσέγγιση σε ό,τι αφορά την τεχνολογική πρόοδο. Με αυτήν την συντονισμένη προσέγγιση μπορούμε να επιτύχουμε συνέργειε και να αποφύγουμε αλληλεπικάλυψη των εργασιών μεταξύ των διάφορων συναρμόδιων αρχών, για παράδειγμα εθνικών αρχών και ε, αρχών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει γενικότερη υποστήριξη για τη δημιουργία μιας ε, γενικότερη δομή στο πλαίσιο τη Ευρωπόλ, η οποία θα ασχολείται ειδικότερα με τι νέε τεχνολογίε, με την ονομασία εργαστήριο καινοτομία. Αυτό το εργαστήριο καινοτομία θα μπορεί να λειτουργήσει ω μια πλατφόρμα ε, μέσω τη οποία θα συνεργάζονται οι διάφορε αρχέ επιβολή τη νομοθεσία και ε, πληροφορική προκειμένου να διευκολυνθεί ο διάλογο μεταξύ του. Και το εν λόγω εργαστήριο θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα μπορούσε να, να παρακολουθεί τις νέες τεχνολογίες, αλλά ταυτόχρονα να αναπτύσσει νέες λύσεις από κοινού με τον κλάδο, πράγμα βέβαια το οποίο μπορεί να δημιουργήσει και σε περισσότερη εξοικονόμηση ε, πόρων σε βάθος χρόνου και να μας καταστήσει και πιο αποτελεσματικούς. Σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά για τη δυνατότητα που μου δώσατε να σας παρουσιάσω αυτά τα στοιχεία ενώπιον της ε, Επιτροπής σας και αναμένω και τις ε, περαιτέρω συζητήσεις μας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη, είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένη για την πρόσκλησή σας και να συμπληρώσω αυτά τα οποία είπε η κυρία Βακούρη για τα θέματα των εσωτερικών υποθέσεων. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το θέμα ασφαλείας, με τα θέματα ασφαλείας και να αναφερθώ σε θέματα τα οποία πραγματικά συμπληρώνουν θα έλεγα αυτά που λέει η συνάδελφος. Εμείς υποστηρίζουμε πλήρως τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της ε, σεξουαλικής βίασης βάρος των παιδιών. Νομίζω ότι έχουμε πετύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα έτσι ώστε να μπορέσουμε να προλαμβάνουμε τέτοιου είδους φρικτά εγκλήματα και τα θύματα φυσικά υπήρξε ομόφωνη θα έλεγα συμφωνία από όλες τις χώρες και ακούσαμε επίσης και από την Ολλανδή Υπουργό στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό στις κάτω χώρες. Να πω ότι ε, στο τέλος αυτής της συνεδρίασης για το συγκεκριμένο θέμα έχει μεγάλη σημασία να έχουμε μια ενιαία φωνή καταδίκης αυτών των εγκλημάτων και επίσης η υιοθέτηση των συμπερασμάτων έγινε με ομόφωνο τρόπο. Από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εμείς εργαζόμαστε για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οδηγίας. Αυτό το οποίο θέλω επίσης να αναφέρω είναι οι συζητήσεις που είχαμε για, την ακροδεξιά, για τον ακροδεξιό εξτρεμισμό στην Ευρώπη. Είναι ένα αναπτυσσόμενο φαινόμενο το οποίο απειλεί τις ευρωπαϊκές αξίες και ως εκ τούτου απαιτεί να υπάρξει μια απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα πρόσφατα γεγονότα στην Γερμανία δυστυχώς επιβεβαίωσαν το χρήσιμο της συζήτησης αυτής και έκαναν ακόμα πιο ξεκάθαρο το ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τις δράσεις μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να σας παρουσιάσω και στα πλαίσια της προσπάθειας να αντιμετωπίσουμε καλύτερα το θέμα των τρομοκρατικών ε, ε, ε, ανακοινώσεων και της δικής της δημοκρατίας στο διαδίκτυο. Θα πρέπει να καταλήξουμε για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου το ταχύτερο δυνατόν. Το άλλο θέμα ασφαλείας το οποίο συζητήσαμε είναι το θέμα της διαλειτουργικότητας διότι αυτό το οποίο χρειαζόμεθα είναι να υπάρξει μια δομημένη αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού από όλα τα κράτη-μέλη και δεν μπορούμε να έχουμε κάποιες χώρες οι οποίες να μένουν πίσω. Ως εκ τούτου λοιπόν, αν ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος καθυστερεί, τότε η ε, σωστή λειτουργία ε, θα απειληθεί. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να στηρίξει τις χώρες που αντιμετωπίζουν θέματα καθυστέρηση και προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με τις χώρες για να προλάβουμε την κατάσταση αυτή. Τέλος, συζητήσαμε την διαλειτουργικότητα των θεμάτων που αφορούν την, ε, την ακτοφυλακή, την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή ενημερώσαμε τα κράτη-μέλη γύρω από αυτό. Έχουμε συγκεκριμένα στάδια και ένα οδικό χάρτη για την πλήρη λειτουργία των θεμάτων της ακτοφυλακής. Για τα θέματα τώρα της μετανάστευσης, εμείς ε, όπως ακριβώς είπε και ο Πρόεδρος, αντιμετωπίσαμε όλους τους, ε, τις οδούς η ελληνική αντιπροσωπεία έθεσε το θέμα της ε, οδού της Ανατολικής Μεσογείου και της αύξησης των αφήξεων τον τελευταίο μήνα. Οι χώρες αναφέρθη, η Ισπανία μάλλον αναφέρθηκε στις δυτικές οδούς για τις ε, ε, εισόδους στην συγκεκριμένη αυτή περιοχή. Η Ιταλία και η Μάλτα αναφέρθηκαν στην κεντρική Μεσόγειο και φυσικά εξετάσαμε και την δήλωση για την έρευνα και αναζήτηση και διάσωση, συγγνώμη, την οποία προώθησε η Μάλτα. Η άποψή μας είναι και το γνωρίζετε αυτό ότι εμείς υποστηρίζουμε σε λειτουργικό επίπεδο εδώ και 1,5 χρόνο τις προσπάθειες ε, και οικονομικά και συντονίσαμε τις ε, ασκήσεις οι οποίες έγιναν για τη διάσωση και έρευνα και γι' αυτό χαιρετίζουμε το επόμενο βήμα θα έλεγα το οποίο αναμένουμε για πιο διαλειτουργικές λύσεις, ολοκληρωμένες λύσεις οι οποίες ε, θα δώσουν πιλωτικά θετικά αποτελέσματα για να καταλήξουμε στη συμφωνία για τη μεταρρύθμιση στον τομέα του ασύλου. Να πω επίσης ότι όλες αυτές οι συζητήσεις για τη μετανάστευση δείχνουν ότι απαιτείται να βρωθούν λύσεις το ταχύτερο δυνατόν. Ε, δεν έχουμε να μιλήσουμε μόνο για μία οδό, εδώ ξέχασα μάλιστα να αναφερθώ και στην Κύπρο. Το θέμα είναι να συζητήσουμε το σύνολο των οδών αυτών και ελπίζω τις επόμενες εβδομάδες ε, να έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη νέα συμφωνία την οποία θα προτείνει η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα της μετανάστευσης προστατεύοντας την καλή δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα μαζί σας. Από πλευράς μου θα ήθελα να σας πω σε προσωπικό επίπεδο ότι έχουμε ένα νέο σκάφος, το Ocean Viking, ε, με χωρητικότητα 176 ατόμων και ε, στα πλαίσια της νέας αυτής δήλωσης θα ξεκινήσουμε τις νέες μορφές συντονισμού για τη σωστή λειτουργία των δράσεων αυτών. Σας ευχαριστώ, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ όλους τους προσκεκλημένους που μίλησαν εκπροσωπώντας την Κομισιόν και το Συμβούλιο για θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Τώρα θα συζητήσουμε μεταξύ μας. Έχουμε ένα πρώτο γύρο με τους συντονιστές. Θα δώσω το λόγο στους συντονιστές που είναι παρόντες. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με την κυρία Μετσόλα και τον κύριο Λέναρτ ως εκπροσώπους του ΕΛΚ. Κυρία Μετσόλα, κάνα δύο λεφτά έχετε στη διάθεσή σας. Σύντομη θα είμαι. Θα ευχαριστήσω τη Φιλανδική Προεδρία για τη δέσμευσή της στον τομέα αυτό και τη Γενική Διευθύντρια για την ενημέρωση που μας έκανε Έχω δύο ερωτήσεις. Μία στην κυρία Στόλα. Αναφερθήκατε στον αριθμό των κρατών μελών που δεν έχουν ε, υποβάλει υποψηφιότητες για τη θέση ε, του εισαγγελέα, του Ευρωπαίου εισαγγελέα, ε, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουν προθεσμία τα κράτη-μέλη. Λίγα είναι αυτά τα κράτη-μέλη και οι προϋποθέσεις που έχουν βάλει οι κυβερνήσεις. Ο λόγος που δεν έχουν ε, προτείνει τους υποψήφιους είναι γνωστός, γιατί έχουν αυτή την υποχρέωση να προτείνουν υποψηφίους. Κυρία Μίχου, για τις συμφωνίες στις οποίες αναφερθήκατε, τη δήλωση που έκαναν κάποια κράτη-μέλη. Από ό,τι ξέρουμε, αυτή η συμφωνία δεν έτυχε επαρκού στήριξη στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Τι σκοπεύει να κάνει η Κομισιόν από εδώ και πέρα, θα προχωρήσει ή θα αντιμετωπίσουμε ακόμη ένα μπλοκάρισμα στο Συμβούλιο και δεν θα μπορέσουμε να απεμπλακούμε από αυτό το πρόβλημα τις επόμενες εβδομάδες. Η κυρία Σίπελ, ένα-δύο λεπτά. Θα μιλήσω γερμανικά. Okay, Ορισμένες φορές διαρωτώμε ε, περί τίνος πρόκειται εδώ, τι ακριβώς συζητούμε. Και διαρωτώμε τι ακριβώς κάνει το Συμβούλιο. Αποφασίζουμε επί νόμων, ε, αποφασίζουμε σε ό,τι αφορά τη συνοριοφυλακή και την ακτοφυλακή. Το Συμβούλιο λέει ότι είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά και στη συνέχεια ε, δεν διασφαλίζει του απαραίτητου πόρου και το ανθρώπινο δυναμικό. Το ίδιο το Συμβούλιο αποφάσισε να ληφθεί η Γενική Εισαγγελία μέσα στην συνθήκη τη Λισαβόνα και ξαφνικά τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να συμμετάσχουν όλα του και εκείνα ε, που συμμετέχουν δεν παρέχουν το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό. Τι να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Έχουμε ένα πακέτο για το άσυλο. Και αναφέρουμε στο πακέτο το οποίο έχει ήδη συμφωνηθεί το οποίο εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν εφαρμόζεται από όλους. Οπότε διαρωτώμε μήπως θα έπρεπε να αξιοποιήσουμε διαφορετικό ε, τρόπο το χρόνο μας. Γιατί τελικά τι κάνουμε εδώ. Αποφασίζουμε κάποιου νόμου, να εγκρίνουμε κάποιου νόμου οι οποίοι τελικά δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Τι είναι όλα αυτά. Αναφερόμαστε για αυξημένου αριθμού ε, αφήξεων ε, στην Ανατολική Μεσόγειο, 11.500 ε, άνθρωποι που καταφθάνουν ε, μηνιαία στην Ελλάδα και μας ανησυχεί αυτό, αλλά δεν μας ανησυχεί το γεγονός ότι ο αριθμός των μεταναστών και των προσφύγων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ μεγαλύτερος σε σύγκριση με αυτόν που καταφθάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούμε ότι οι τελευταίες εξελίξεις θα μπορούσαν να συμβάλλουν ε, στην αύξηση του αριθμού των αφήξεων. Αλλά ας αναφέρουμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η Τουρκία λοιπόν έχει ξεκινήσει εμπόλεμη σύραξη στη Συρία μια, ένας πόλεμος ο οποίος δεν έχει ανακοινωθεί ε, επισήμως. Αλλά όταν υπάρχει στρατιωτικού χαρακτήρα επίθεση από τη μία χώρα εις βάρος μιας άλλης προκειμένου να προστατεύσει τα ε, γεωπολιτικά της συμφέροντα ή ε, επειδή υπάρχει μια νεύρωση από την πλευρά εκείνης της χώρας ό,τι αφορά μια εθνική μειονότητα με την ονομασία Κούρδη, τότε τι άλλο και εμεί τι λέμε από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να δώσουμε περιττέρω και άλλα χρήματα στην Τουρκία. Και θέτω και πάλι ένα ερώτημα για το οποίο ποτέ δεν έλαβα κάποια απάντηση. Σε τι ακριβώ χρησιμεύει, πώ αξιοποιούνται αυτοί οι πόροι του οποίου παρέχουμε στην Τουρκία. Πραγματικά είναι προ ε, όφελο των προσφύγων ή αξιοποιούνται για διαφορετικού σκοπού. Και ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα να κάνω σε ό,τι αφορά τους σε ε, τι νέε επιθέσει, τη ρητορική μίσου και τη διάδοσή τη και ούτω καθεξής. Ναι, είναι τρομακτικά όλα αυτά επειδή εξαπλώνεται τόσο πολύ ρητορική μίσου. Αλλά ορισμένε φορέ ε, διαρωτώ με γιατί αναφερόμαστε τόσο στη ρητορική μίσου και στην παραπληροφόρηση στον κυβερνοχώρο ε, αλλά ταυτόχρονα δεν αναφερόμαστε στα όσα συμβαίνουν στην πραγματική ζωή. Βλέπουμε δηλαδή το πώς, ε, τι συμβαίνει από την πλευρά ε, και για παράδειγμα των ιερωμένων για παράδειγμα, και των εκπροσώπων τη Εκκλησίας όπως είδαμε και στο πλαίσιο ε, του πρόσφατου διορισμού στην ε, Πολωνία ε, και σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την, και την προστασία των παιδιών. Ναι, είναι όλα αυτά σοβαρά αλλά από την άλλη πλευρά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί ε, δεν ανησυχούμε σε ό,τι αφορά τα πραγματικά προβλήματα που λαμβάνουν χώρε στι γειτονικέ μα χώρε και μα ανησυχούν όλα τα υπόλοιπα στον κυβερνό χώρο. Renew, Intveld. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ του τέσσερι ομιλητέ για τι παρεμβάσει του. Πριν να υποβάλω τι ερωτήσει μου, μία ερώτηση προ εσά, Πρόεδρε, για τον τρόπο που συνεδριάζουμε εδώ. Υποτιθέτω ότι γίνεται εδώ μια πολιτική λογοδοσία, ένας πολιτικός διάλογος ε, οι πολιτικοί που είναι υπεύθυνοι έρχονται εδώ και μιλούν, καταθέτουν. Με κάθε σεβασμό που έχω και εκτίμηση προς τις τέσσερις ομιλήτριες, νομίζω ότι θα πρέπει να εκπροσωπείτε το πολιτικό επίπεδο, γιατί εσείς δεν μπορείτε να μας δώσετε πολιτικές απαντήσεις. Τώρα για τα θέματα τα οποία συζητούμε, θα κάνω μια επιλογή, γιατί ακούστηκαν πολλά για το γραφείο του, της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, μία από τις ανησυχίες μου είναι ότι υπάρχει σημαντική αντίθεση προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ακόμα, και θα ήθελα να δοθούν επαρκή μέσα και υποστήριξη ήδη στη φάση εδώ τη σύστασή τη της Ευρωπαϊκής εισαγγελία και από το Συμβούλιο και από την Κομισιόν και από το Κοινοβούλιο. Τι άποψη έχετε επίσης. Τα μέλη του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δηλαδή το να διορίζει ένα κράτος μέλος, έναν εισαγγελία προϋπόθεση για να παίρνει ε, χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Επίσης, για τη λήψη ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων. Είναι πολύ πρόωρο αυτό το θέμα. Είναι απαράδεκτο που τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών τα διαπραγματευόμαστε και τα απεμπολούν οι γραφειοκράτες και κλεισμένων των θυρών. Ε, με εκνευρίζει πάρα πολύ το γεγονό ότι δεν λάβατε καθόλου υπόψη στην γνωμοδότηση για τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασία Δεδομένων. Επίση, θα ήθελα να μου πείτε λιγάκι την άλλη σύμβαση που διαπραγματεύεται και κλεισμένων των θυρών τη Βουδαπέστη για το κυβερνοέγκλημα. Προχωράτε πολύ γρήγορα στι διαπραγματεύσει ε, αυτών των συμφωνιών ε, ή στην πρόθεση νομοθεσίε, αλλά δεν υπάρχουν οι απαραίτητε νομικές ασφαλιστικές δικλείδες. Π.χ. η οδηγία για την ε, εφαρμογή του νόμου για την προστασία των δεδομένων έχει εφαρμοστεί από 20 κράτη-μέλη μέχρι στιγμής. Αυτό σημαίνει ότι 8 κράτη-μέλη προσπαθούν, λειτουργούν μάλλον με το, με το πλαίσιο του 2008. Την απόφαση πλαίσιο. Αυτό είναι γελίο. Θα πρέπει να υπάρξει πρόταση της Κομισιόν για κανονισμό για να αντικαταστήσουμε την οδηγία αυτή. Επίσης, για την έρευνα και διάσωση και το θέμα των προσφύγων. Δεν ξέρω τι να πω. Ακούω τη Φιλανδική Προεδρία που μιλάει για την αύξηση τη βοήθεια και τη συνεργασία προ την Τουρκία. Τι να πω γι' αυτό. Η Τουρκία ξεκινάει ένα πόλεμο. Θέλει να στείλει πίσω 2 εκατομμύρια πρόσφυγες στην Συρία, ετοιμάζουν και εθνική κάθαρση και εμεί θέλουμε να αυξήσουμε τη βοήθεια και τη συνεργασία με την Τουρκία. Σαν να ζούμε σε διαφορετικού πλανήτε είμαστε. Αυτή η δήλωση για την Τουρκία δεν θα πρέπει να υπάρχει καν. Ο κ. Ερντοάν μα ε, ε, εκβιάζει κιόλα. Είμαστε ανοιχτοί στον εκβιασμό του. Εμεί δεν ξέρουμε να απαντήσουμε. Και μιλάμε για βοήθεια και συνεργασία. Είναι λάθο αυτό. Και ένα τελευταίο ερώτημα, Πρόεδρε. Για αυτέ τι πληροφορίε. Ε, υπάρχει την, ε, το ψήφισμα τη περασμένη εβδομάδα που υιοθετήσαμε. Και χθε, μετά τα αποτελέσματα των πολωνικών εκλογών βλέπουμε ότι ο, ο διευθυντής της ε, κρατικής πολωνικής τηλεόρασης ήταν παρόν ε, τη μέρα των εκλογών ε, ως εκπρόσωπος ε, του κυβερνητικού κόμματος. Ναι, ναι, κλείνω. Πώς δεν κάνει τίποτα η Κομισιόν για αυτές τις πληροφορίες που διαδίδουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Αυτά είναι προς το Συμβούλιο, από τους α, ε, πράσινους. Ούτε ο κύριος Ρένκελ, ούτε ο κύριος Τρίνκ είναι παρόντες εδώ. Είπαν ότι δεν θα έρθουν, έχουν κάποιο, κάποια ανηλυμένη υποχρέωση εκτός Κοινοβουλίου. Ο κύριος Προκατσίνη δεν είναι εδώ. Άρα μπορούμε να δώσουμε το λόγο στην κυρία Ταρντίνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για το θέμα της μετανάστευσης. Σας παραπέμπω σε αυτά που είπε ο συνάδελφος ή συνάδελφος για τη συνεργασία με την Τουρκία. Γιατί μας εκπλήσει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, την ιστορική στιγμή, η Ευρώπη σκέφτεται έστω να μιλάει για συνεργασία με την Τουρκία. Επίσης, γίνονται διαδηλώσεις για τη συμφωνία με την Μάλτα, που παρουσιάζεται ως μεγάλη συμφωνία. Να υπενθυμίσουμε ότι όχι μόνο ε, επικυρώθηκε από τέσσερα κράτη-μέλη, αλλά άλλα τρία κράτη-μέλη που δεν είναι σημαντικά για την ε, επίτευξη πλειοψηφίας, ε, είπαν ότι είναι διατεθειμένα να προσχωρήσουν αυτή τη συμφωνία. Υπάρχει μια κατάσταση, ένα κράτος που λέει ότι πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί περισσότερα, χωρίς να προτείνει τίποτα όμως. Ε, κάποιο άλλο κράτος που έκανε, υποτίθεται, πάρα πολλές ε, προσπάθειες για να στηρίξει τη Συμφωνία της Μάλτας για ένα συστηματικό καταμερισμό των ε, μεταναστών. Ποια είναι η μεγάλη επιτυχία για τη Συμφωνία της Μάλτας. Ε, το παρουσιάζεται ως πιλωτικό πρόγραμμα. Νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια με τέτοια εντυπωσιακά προβλήματα που έχουμε, μιλάμε απλώς για πιλωτικά προγράμματα. Δεν θέλουμε ad hoc λύσεις για κάθε αποβίβαση από σκάφη. Θέλουμε αποτελεσματική διαχείριση ενός φαινομένου που έχει κολοσιαίε διαστάσεις. Ποια είναι η λύση που προτείνει η Ευρώπη. Το ρωτάω ακόμα μια φορά. Ίσως να αφήσουμε μόνα τους τα κράτη τα οποία είναι τα κράτη της πρώτης υποδοχής. Μιλάτε για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία. Και εντός παρενθέσεως και παρόδο μόνο μιλάτε για την Ιταλία. Ε, τι απαντήσεις θα δώσει η Ιταλία στους πολίτες. Για την Ιταλία και τη Μάλτα. Το θέμα της αναδιανομής σε θελοντική βάση, όπως προβλέπει η Συμφωνία της Μάλτας, αφορά τα άτομα τα οποία αποβιβάζονται από σκάφη ΜΚΟ, μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ξέρουμε όμω ότι οι περισσότερε αυξήσει δεν φτάνουν με αυτά τα σκάφη, αλλά φτάνουν με ιδιωτικά σκάφη. Δεν, φτάνουν δηλαδή με σκάφη των κοιό. Ελπίζω να μα δοθεί κάποτε μία απάντηση. Τι σκοπεύει να κάνει η Ευρώπη για αυτό το πρόβλημα. Ernst ε, δεν ήταν εδώ, αλλά τώρα κατέφθασε στην αίθουσα, οπότε μπορείτε να πάρετε το λόγο, κυρία Ernst, αν επιθυμείτε. Έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων την οποία διεξάγουμε ε, με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σε ό,τι αφορά τι εσωτερικέ επιθέσει και τη δικαιοσύνη, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα τελευταία συμπεράσματα του Συμβούλου. Παρακαλώ, κυρία Ένστε. Ναι, ε, δυστυχώ αγαπητοί συνάδελφοι, μερικέ φορές καταφθάνουμε αργοπορημένοι έτσι, γιατί ε, δεν είναι εύκολα τα πράγματα σε ό,τι αφορά την κίνηση, ειδικότερα τη Δευτέρα το απόγευμα. Λοιπόν, θέλω να θέσω κάποια ερωτήματα. Καταρχήν, Μόρια. Τι σκοπεύει να κάνει η Επιτροπή και το Συμβούλιο προκειμένου να βελτιωθούν εκεί τα πράγματα Υπάρχουν δηλαδή κάποια σχέδια προκειμένου να γίνει ανακατανομή εκεί των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί, ε, όχι μόνο εντό τη Ελλάδα αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη, γιατί πραγματικά διαβιώνουν υπό καταστροφικέ ε, συνθήκε. Τώρα, δεύτερο ζήτημα. Έχουμε έναν πόλεμο ο οποίο ε, διεξάγεται στα βόρεια τη ε, Συρία ε, και αρχίζουν να κατευθύνονται όλοι αυτοί οι πρόσφυγε 200.000 άτομα προ τα εσωτερικά τη Συρία, αλλά δεν ξέρουμε πώ τα προ τα που θα συνεχίσουν να κατευθύνονται, αν θα υπάρξουν δηλαδή νέε μεταναστευτικέ οδοί που θα υπάρχουν. Και σίγουρα το γεγονό ότι τώρα θα υπάρξουν κάποιοι μαχητέ ε, του Άσις που θα ενεργοποιηθούν και πάλι θα δημιουργήσει επιπλοκέ. Οπότε ρωτώ την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ε, είναι διατεθειμένοι να συνεχίσουν ε, με αυτό το ορθόδοξο δόγμα τους ή θέλουν, ε, για παράδειγμα, ε, να σταματήσουν να εφαρμόσουν αυτή τη συμφωνία συνεργασία ε, με την Τουρκία. Προκειμένου δηλαδή να μην επιτρέπουν στην Τουρκία να του εκβιάζει σε ό,τι αφορά δηλαδή την αποδοχή προσφύγων. Γιατί πραγματικά η λόγω συμφωνία, κατά τη δική μου άποψη, δεν λειτουργεί και πραγματικά ουσιαστικά αποτελεί το προϊόν εκβιασμού από την πλευρά τη Τουρκία και είναι ντροπή για του Ευρωπαίου πολίτε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Α ε, κάνουμε τώρα ένα πρώτο γύρο ερωταπαντήσεων πολύ γρήγορα, αν ε, έχετε λίγο χρόνο. Λοιπόν, τρία λεπτά ο καθένα από του ομιλητέ εδώ του πάνελ, γιατί υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι ακόμα που θα ήθελα να παρέμβω. Α προβλέψουμε λοιπόν 20 ακόμα λεπτά ε, για το εν λόγω ζήτημα στην μερίσια διάταξή μας. Οπότε παρακαλώ, ομιλητέ εδώ του πάνελ, τρία λεπτά καθένας. Η ε, κυρία Αστολά, καταρχήν σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, να κάνω κάποια σχόλια. Σε ό,τι αφορά την Εισαγγελία, καταρχήν, και εδώ αναφέρομαι και στο ζήτημα και στο ερώτημα του κατά πόσο έχει νόημα του να εγκρίνουμε νέα νομοθεσία όταν η φυστάμενη νομοθεσία δεν εφαρμόζεται. Να πω ότι σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση, δηλαδή το χρονοδιάγραμμα έχει προβλέψει τη δημιουργία της έως τα τέλη του 2020 και επιχαίρω ιδιαίτερα το γεγονό ότι ε, αποφασίσαμε σε ό,τι αφορά το διορισμό του Αρχή Εισαγγελέα γιατί με αυτόν τον τρόπο θα ξεκινήσουν να κινούνται τα πράγματα. Τώρα σε ό,τι αφορά ε, κάποιου ε, διορισμού, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα γίνει, σε ό,τι αφορά δηλαδή, τους υποψηφίου από την πλευρά ε, Το αρχικό χρονοδιάγραμμα ήταν τέλη Μαρτίου. Αλλά ο Πέτροπος ε, τώρα έχει αξιώσει ιδιαίτερα εμφατικά τον διορισμό αυτών των υποψηφίων από την πλευρά των κρατών ε, μελών, δηλαδή από το Συμβούλιο. Οπότε παρότι δεν έχει οριστεί ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, νομίζω πω έχει περάσει αυτό το μήνυμα, ότι είναι επιτακτική ανάγκη δηλαδή να διοριστούν και οι υπόλοιποι εισαγγελεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που αναφέρθηκε, ότι υπάρχουν δηλαδή αντιρρήσει ό,τι αφορά τη δημιουργία τη ίδια τη εισαγγελία από την πλευρά των κρατών μελών. Εμεί ε, χαιρόμαστε ιδιαίτερα για το γεγονό ότι υπάρχουν τόσα πολλά κράτη-μέλη που ήδη συμμετέχουν και η Σουηδία, για παράδειγμα, σε λίγο θα ε, συμπεριλαμβάνεται σε αυτά τα κρατη που συμμετέχουν. Οπότε πραγματικά έχει γίνει πολλή δουλειά από τότε που ξεκινήσαμε και εν λόγω εισαγγελία θα μπορέσει να παίξει ένα ισχυρό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά του ε, πόρου και τη διάθεσή του, ναι, πράγματι εδώ ε, αυτό θα πρέπει να το κινήσουν, να το προωθήσουν τα ίδια τα κράτη-μέλη, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ανησυχώ ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την έλλειψη πόρων της εισαγγελίας. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά το να καταστεί ω προπόθεση κάτι τέτοιο για την εκταμίαση ε, κοντιλιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω γνωρίζετε συζητούμε αυτή την περίοδο ε, το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο και εκεί ακριβώ γίνεται λόγο ε, και για την τήρηση του κράτου δικαίου. Και δηλαδή το πώ τελικά γίνεται η εκταμίαση αυτών των κοντιλιών και δαπάνη τους. Αλλά αυτό θα το δούμε και αργότερα. Τώρα σε ό,τι αφορά τη σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ, θεωρήθηκε πως είναι πολύ πρόημο κάτι τέτοιο, μια τέτοια συμφωνία δηλαδή, γιατί και γίνεται και κλεισμένο των θηρόν συζήτηση και δεν υπάρχουν και δικλείδες ασφαλείας. Και ήταν ξεκάθαρο στην εντολή ότι η Επιτροπή δεσμεύεται από τον τρόπο που κινούνται οι συζητήσει σε ό,τι αφορά το ζήτημα τη ε, συγκέντρωση των ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων και στο πλαίσιο δηλαδή και τη διαπραγμάτευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. κύριο Ζέντερ, που είναι ο νέο ε, επίτροπο, το κατέστησε και από τη δική του πλευρά αυτό πολύ σαφέ, ότι δηλαδή εξαρτώμαστε στην εντολή μα από πλευρά τη Επιτροπή από τι διαπραγματεύσει που τρέχουν και με, την, ε, με το Κοινοβούλιο. Κυρία Βακούρη, για τα θέματα ε, εσωτερικών υποθέσεων. Όχι δικαιοσύνη, διορθώνει ο πρόεδρο. Θέλετε να προσθέσετε κάτι. Άκουσα μία-δύο ερωτήσει για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εξήγησα τα θέματα χρηματοδότησης και τα του διορισμού των Ευρωπαίων ε, εισαγγελέων. Το Συμβούλιο είναι έτοιμο να προβεί στους διορισμούς των Ευρωπαίων εισαγγελέων, των μελών δηλαδή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η κυρία Βακούρη τώρα για τα θέματα εσωτερικών υποθέσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα περισσότερα θέματα, τα περισσότερα ερωτήματα που ακούστηκαν από τους βουλευτές για ζητήματα εσωτερικών υποθέσεων αφορούσε τη μετανάστευση. Θα ήθελα να απαντήσω για αυτά. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Μίχου, η οποία θα συμπληρώσει τα όσα θα πω εγώ. Πιστεύουμε ότι είναι ευθύνη της Προεδρίας να εξασφαλίσει ότι Κανένα κράτος μέλος το οποίο δέχεται πίεση, μεταναστευτική πίεση, δεν μένει μόνο του. Αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις οδούς στη Μεσόγειο, στη συζήτηση που έγινε στο Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα. Σε αυτή τη φάση φαίνεται σαφές ότι έχουμε διαφορετικές οδούς και επομένως δεν μπορούμε να βρούμε μία και μόνη λύση για κάθε οδό. Μία λύση για όλες τις οδούς. Συγγνώμη. Η Ιταλία, Μάλτα, η Γαλλία και η Γερμανία είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα πιλωτικά τους προγράμματα και την εφαρμογή του πιλωτικού συγγνώμη, προγράμματος. Ένα είναι το πρόγραμμα που ε, είναι και ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να το προωθήσει. Για τη βοήθεια που δίδεται στα κράτη-μέλη, όπως είπα και στην αρχική μου ομιλία, η Κομισιόν και οι διάφοροι οργανισμοί ετοιμάζουν νέους τρόπους για να δώσουν περαιτέρω βοήθεια. Αυτό το ξεκαθάρισε η Κομισιόν και στο Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα. Τώρα, για την κατάσταση εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως πέρα από τα νότιο-ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνω τις επικρίσεις, η κατάσταση είναι ανησυχητική. Και ακριβώς γι' αυτό η Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αντιμετωπίσει και θα συζητήσει αυτό το θέμα αυτή τη βδομάδα. Οι Υπουργοί Εσωτερικών θα παίξουν το ρόλο τους όταν μιλάμε για συνεργασία με μη ενωσιακές χώρες παίζουν και αυτοί κάποιο ρόλο. Θα πρέπει να περιμένουμε όμως τις συζητήσεις πρώτα που θα κάνουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η Κομισιόν θα πει και άλλα πράγματα από αυτού του θέματο. θέματος. Έχουμε κάποια σχέδια για έκτακτες υποθέσεις και αυτά ακριβώς είναι ευθύνη των Υπουργών Εσωτερικών. Η κυρία Μίχου, για συμπληρωματικά σχόλια. Θα ξεκινήσω με το θέμα έρευνας και διάσωσης. Έχουμε τις τέσσερις χώρες, Ιταλία, Μάλτα, Γερμανία και Γαλλία και διάφορα άλλα κράτη-μέλη, τα οποία είπαν ξεκάθαρα ότι θα συμμετάσχουν και θα υποστηρίξουν την προσπάθεια. Έχουμε διάφορα κράτη-μέλη που είπαν ότι εξετάζουν θετικά το θέμα αυτό και θα το αξιολογήσουν και θα απαντήσουν. Όλα όμως είπαν ότι περιμένουν να βρεθεί ευρωπαϊκή λύση για τη μεταρρύθμιση του ασύλου και έχουμε και κάποια κράτη-μέλη τα οποία έχουν θέσει κάποια προβλήματα για το κατά πόσον ε, προσκαλούμε περισσότερους μετανάστες μια τέτοια δήλωση. Η δήλωση ως έχει, έχει κάποια στοιχεία λειτουργικά που τα είδαν η Κομισιόν, τα κράτη-μέλη, η Ιταλία και η Μάλτα και όσοι ασχολούνται με, την κατάσταση ήδη από πέρυσι. Πέρυσι, ε, μάλλον την Παρασκευή, έγινε μια συνάντηση για τις, την κλασική διαδικασία λειτουργίας για το πώς διεξάγονται στη Μάλτα και στην Ιταλία αυτές οι επιχειρήσεις. Ποιος θα βοηθήσει, τι θα δώσει η ΕΑΣΟ, η BCG, η Europol, η Κομισιόν και για το θέμα του χρονοδιαγράμματος, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι μέσα σε ένα μήνα όλοι όσοι είναι τούντες άσυλου θα πρέπει να μετεγκατασταθούν. Είδαμε κάποιες καθυστερήσεις σε θέματα μετεγκατάστασης. Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα, το είπα και στην αρχή. Με βάση την εμπειρία που θα συλλέξουμε και θα αποκτήσουμε, θα φτιάξουμε μία πιο μόνιμη λύση. Αυτή δεν είναι η μόνιμη λύση. Βοηθάει τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια να δουν ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους. Είναι ένα θετικό βήμα προς την εξέβρεση μιας πιο μόνιμης λύσης. Για την Τουρκία. Τα λεφτά που δίνουμε στην Τουρκία δίνονται για τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Για δασκάλους στα σχολεία, για τρόφιμα. Γι' αυτό ακριβώ παραπονιέται η Τουρκία ότι δεν προχωράμε γρήγορα. Γιατί πληρώνουμε μηνιαία τα ποσά αυτά. Έχουμε δεσμεύσει τα λεφτά αυτά, αλλά δεν τα δίνουμε στην Τουρκία. Γιατί έχουμε όλα μαζί, γιατί έχουμε αυτές τις καθυστερήσεις. Συνεχίζουμε, λοιπόν, Και την περασμένη εβδομάδα έγινε συζήτηση και εν συνεχεία η Κομισιόν δημοσίευσε τα σχετικά στοιχεία της συζήτησης για το τι πληρώνουμε ακριβώς στην Τουρκία. Προχωρούμε λοιπόν με αυτή τη συνεργασία. Τώρα Βεβαίω, τα ποια είναι τα επόμενα βήματα, αυτή είναι πολιτική υπόθεση και το συζητούν οι Υπουργοί Εξωτερικών καθώς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα συζητήσουν την κατάσταση στη Συρία και τις δράσεις και τη στάση της Τουρκίας, ε, την οποία καταδικάζουν όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, για την Ελλάδα. Οι συνάδελφοι είπαν, οι βουλευτές είπαν, ότι μιλήσαμε μόνο για το πώς βοηθάμε την Ελλάδα για τη Μόρια. Υπάρχουν διμερείς συμφωνίες με κρατημέλη για τους ασυνόδευτους ανήλικους και για το πώς θα πάρουμε κάποιους ασυνόδευτους ανήλικους που έχουν μετεγκατασταθεί εντός της Ελλάδας. Χρηματοδοτούμε περισσότερο ε, για να μεταφερθούν άνθρωποι σε ευάλωτη κατάσταση από τα νησιά στην ενδοχώρα της Ελλάδας. Θέλουμε τώρα να βρούμε πιο βιώσιμες λύσεις. Υπάρχουν ε, σχέδια ε, στην Ελλάδα για τη μεταρρύθμιση του εθνικού καθεστώτος ασύλου καθώς και για πιο μόνιμες λύσεις ε, κατάσταση στην ενδοχώρα και πιο μόνιμες λύσεις ε, στα νησιά. Στην Κομισιόν έχουμε σχέδια κατεπήγοντος σε περίπτωση που συμβεί κάτι τις επόμενες εβδομάδες. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι τεχνικός πώς όλοι οι οργανισμοί και οι υπηρεσίες μας έχουν ετοιμαστεί μετά από συζήτηση με τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο για διάφορα σενάρια που μπορεί να ανακύψουν τις επόμενες εβδομάδες και η Europol, καθώς και η Frontex και η BCG. Εξετάζει τα σημεία εισόδου για να υπάρχει περισσότερη περισσότερη έλεγχη και καταγραφή και στην Ελλάδα και στην Ιταλία και στην Κύπρο και στη Μάλτα και στην Ισπανία. Εξετάζουμε όλες τις οδούς λοιπόν. Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα. Μαζί πρέπει να βρούμε μόνιμες λύσεις. Ετοιμαζόμαστε, ελπίζω να μας βοηθήσετε να τις βρούμε. είτε να μονιμοποιήσουμε τις λύσεις που έχουμε επιτάπητος ή οποιασδήποτε άλλες λύσεις βρούμε, αλλά ό,τι βρούμε θα το συζητήσουμε μαζί σας. Τίνω να υπάρξει ένας δεύτερος γύρος, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε ξεπεράσει το χρόνο και έχουμε και άλλα θέματα. Και γι' αυτό θα, θα δώσω το λόγο σε αυτούς που τον επιθυμούν, αλλά όχι πάνω από ένα λεπτό καθένας, για να μπορέσουμε να καλύψουμε την καθυστέρηση. Μωράες, έχετε το λόγο. Για τη Μόρια και για την έρευνα και διάσωση. Άκουσα γι' αυτά και γι' αυτό θα αναφερθώ αποκλειστικά στην οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Δεν ξέρω αν θα συζητηθεί ε, την επόμενη συνάντηση των Υπουργών σε 10 μέρες. Εμείς την επόμενη εβδομάδα θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό στην Ολομέλεια. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν τι γίνεται με το Συμβούλιο Υπουργών. Οι συνάδελφοι έθεσαν τις ερωτήσεις για τη Μόρια και άλλα θέματα. Ευχαριστώ κύριε Μωράες Γεζόφσκι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρέπει να είσαστε πολύ αυστηροί και για τους συντονιστές. Μία απλή ερώτηση θέλω να θέσω. Εμείς ε, δίνουμε αγώνα για τη δημοκρατία. Και πριν ένα χρόνο άλλαξε το καθεστώς της Μαλδίβες. Οι Μαλδίβες είναι μια μικρή χώρα, νησιωτική, χίλια νησιά, στον Ινδικό ωκεανό. Και ζητούν οι Μαλβίδες ε, ε, απελευθέρωση στο καθεστώς χορήγησης θεωρήσεων. Τι σκοπεύετε να κάνετε για αυτή τη μικρή και όμορφη χώρα η οποία ε, μας υποστηρίζει στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Thank you, Mr. Chair. Mm, uh, after... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά από αυτά που είπατε για την εισβολή στη Συρία από την Τουρκία, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι δύσκολο να συζητήσουμε όλα τα υπόλοιπα θέματα. Ε, το θέμα της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση, προφανώς αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό και θα ήθελα να ρωτήσω τι συγκεκριμένες δράσεις θα αναλάβει το Συμβούλιο τις επόμενες εβδομάδες για τις διαπραγματεύσεις γύρω από το θέμα αυτό. Ο κύριος Μορένο Σάντσες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα. Η κυρία Μίχου και άλλοι μας είπαν για τα θέματα των αφήξεων των μεταναστών είναι κάτι το οποίο ε, μας απασχολεί και είναι κατεπήγον. Εγώ πριν 15 χρόνια ήμουν εθνικός βουλευτής και τότε ήταν κατεπήγον και πάρα πολλές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ε, έχουν ληφθεί μέχρι τώρα, από τότε όπως τα Σέγγεν, αλλά το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, σε τι χρονισμό θα έλεγα θα γίνουν τα βήματα αυτά. Και επίσης θα ήθελα να μάθω τι θα γίνει και με το θέμα των μη συνοδευομένων ανηλίκων. Πότε θα έχουμε επιτέλους μια ενιαία στάση γύρω από αυτό. Ο κύριος Ούρλιχ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αναφερθήκατε και στην καταπολέμηση της ακροδεξιάς λευκής λεγόμενης τρομοκρατίας όταν κάποιος είναι εξτρεμιστής φυσικά αλλά δεν αναφερθήκατε στον Ισλαμιστικό εξτρεμισμό γιατί και αυτός αποτελεί μια πάρα πολύ σημαντική και επίσης η καταπολέμηση των κομμουνιστών της νέας γενεάς, οι οποίοι ζητούν για την απεριόριστη ισότητα, όχι ισότητα ευκαιριών, αλλά άλλες ύποπτες πλευρές. Πολύ επικίνδυνο αυτό για την κοινωνία. Ο εξτρεμισμός, ο θρησκευτικό, ο πολιτικός, της δεξιάς, της αριστεράς, όλα αυτά είναι επικίνδυνα. Τα αγνοείτε. Ο κύριος Βαντερντρίσε. για αυτά τα οποία είπε η κυρία Μίχου σε σχέση με την ακροδεξιά τρομοκρατία και για την ρητορική μίσους η οποία αυξάνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μας ενδιαφέρει και στο Βέλγιο στα πλαίσια των στοιχείων της εθνικής ασφάλειας. Υπάρχουν, υπάρχει κατάλογος, ε, ε, θα έλεγα υπόπτων και κάποιοι από αυτούς, ένας μικρός αριθμός είναι έτοιμος να προβεί σε βίες ενέργειες και στις κάτω χώρες ε, με βάση τα στοιχεία της Εθνικής Ασφάλειας το 2018 η άκρα αριστερά απεδείχθη πιο βίαιη από την άκρα δεξιά. Ε, στην Ιταλία είχαμε ενέργειες τρομοκρατικές και επιθέσεις εις βάρος της Λίγκα, εις βάρος των υποψηφίων της AFD στην Γερμανία. Ε, δεκάδες χιλιάδες εξτρεμιστές της αριστεράς δρούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε ποιες είναι οι προτεραιότητές σας, δεν αναφερθήκατε σε αυτούς τους εξτρεμιστές της αριστεράς είναι θέμα προσανατολισμού, αυτό οφείλεται στον τρόπο που υπολογίζεται τα πράγματα, υπολογίζεται τον κίνδυνο εις βάρος των κοινωνιών μας. Να πω επίσης ότι το Συνδικάτο των Αστυνομικών ζήτησε σήμερα στο Βέλγιο να διαπιστωθεί ότι θα πρέπει να ληφθούν εις βάρος των οργανώσεων της δεξιάς μέτρα που δεν έχουν ληφθεί εις βάρος των οργανώσεων της αριστεράς. Λοιπόν, πρώτα θα ακούσουμε τα θέματα της δικαιοσύνης και μετά τα θέματα των εσωτερικών υποθέσεων. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Ναι, νομίζω πως έγινε, τέθηκε ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά την ισότιμη μεταχείριση. Ένα θέμα το οποίο ε, υπάρχει εδώ και πολύ καιρό. Αυτό που θα κάνουμε από την πλευρά του, της θα γίνει ε, μια συζήτηση πολιτικής στο Συμβούλιο ε, ΕΠΣΚΟ στις 24 ε, Οκτωβρίου προκειμένου να προσπαθήσουμε να βρούμε κάτι ανάλογο ή κάτι το οποίο να μας επιτρέψει να σημειώσουμε κάποια πρόοδο. Παρακαλώ, Ο τη Γενική Διεύθυνση. Κυρία Στόλα. όπως αναφέρθηκε και από την υποψηφία πρόεδρο, θα περιμένει καταρχήν να δει το τι θα συμβεί ε, σε επίπεδο Συμβουλίου ΕΠΣΚΟ και μετά θα δει πώς θα κινήσει τα πράγματα περαιτέρω. Σε ό,τι αφορά τώρα τις συμπληρωματικές ε, ε, οδηγίες, σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της σύμβασης, νομίζω και εδώ τα πράγματα βρίσκονται στα χέρια του Συμβουλίου, δηλαδή το πώς θέλει να δώσει συνέχεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη ρητορική των εξτρεμιστών, ο κώδικας διοντολογία που υφίσταται φυσικά ε, είναι κατά όλων των ειδών τη ρητορικής ε, μίσους ε, από οποιαδήποτε πηγή και προέρχεται αυτή η ρητορική μίσου, αλλά όπω είπα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τώρα νέε προκλήσει. Και μία από αυτέ τι νέε προκλήσει είναι εκείνη η οποία γενικά επιδίδονται στη ρητορική μίσου και ε, η σύνδεσή τους όπως είπαμε με αυτούς που είναι ακριβώς ακραίων πεπιθήσεων. Αλλά κατά την δική μας άποψη είναι ξεκάθαρο στο κώδικα θεωτολογίας ότι με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίσουμε κάθε είδους ρητορική μίσους. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τώρα τις, τις εσωτερικές υποθέσεις. Ναι, απαντώ. Σε ό,τι αφορά τον βίο η Προεδρία υπογράμμισε την ανάγκη του αντιμετωπίσουμε και πολιτικά και, και, και πολιτική και ιδεολογική ε, ρητορική και εξτρεμισμό και ε, όπως γνωρίζετε εδώ και πολύ καιρό εδώ και κάποια χρόνια ε, πάντοτε δίναμε περισσότερη έμφαση στους τζιχαντιστές και τον βίο εξτρεμισμό τους. Ε, ταυτόχρονα διαπιστώνουμε ότι με βάση τις πιο πρόσφατες εκθέσεις ο βίος εξτρεμισμός της ακροδεξιάς αυξάνεται και αυτό βέβαια είναι ένα ανησυχητικό φαινόμενο και γι' αυτό το λόγο στο τελευταίο συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας δηλαδή δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση ακριβώς σε αυτό το ζήτημα δηλαδή του ακροδεξιού βίου εξτρεμισμού. Αλλά ταυτόχρονα θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι δεν είναι ε, ο στόχος ε, της Προεδρίας να εστιάζουμε μόνο σε επιμέρους πτυχές αυτού του φαινομένου. Θέλουμε να το, επι... να το αντιμετωπίσουμε σε όλα τα επίπεδα και με όλες τις μορφές. Ναι, η κυρία Μίχο έχει το λόγο. Ναι, ε, πολύ συγκεκριμένα θα απαντήσω σε ένα ζήτημα σε ό,τι αφορά την πολιτική μας για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Υπάρχει ήδη καταρχήν μια οδηγία που ισχύει και με βάση την οποία μπορούμε να κινηθούμε. Αλλά μία από τις ε, προτεραιότητες μας είναι το να κάνουμε ακόμα περισσότερες προσπάθειες εδώ, ε, προκειμένου όχι μόνο να εφαρμόζεται και να επιβάλλεται αλλά και προκειμένου να αντιμετωπίσουμε οποιασδήποτε ελλείψεις. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι εργαζόμαστε σκληρά και αναμένουμε τον διορισμό της Νέας Επιτροπής. Και από αυτά που ακούμε και από αυτά που βλέπουμε, μέχρι τα τέλη του έτους θα γνωρίζουμε ακριβώς όποιο θα είναι το μέλλον. Σε ό,τι αφορά τώρα την πολιτική θεωρήσεων, όπως γνωρίζετε, έχουμε μια διαφορετική πολιτική για ένα διαφορετικό προσανατολισμό τώρα, αλλά εξετάζουμε αυτή την περίοδο ε, ορισμένες χώρες, ανά περίπτωση, την κάθε μία δηλαδή ξεχωριστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ για την προσπάθεια που κάνατε εδώ να δώσετε πολύ σύντομε απαντήσει, ε, παρότι τέθηκαν πολλά ερωτήματα προς σα. Ευχαριστούμε λοιπόν όλους εδώ τους καλεσμένους μας, ε, τους ομιλητές, ε, τόσο από την πλευρά του Συμβουλίου και τη Προεδρία, και από την πλευρά της Επιτροπής, από την πλευρά των δύο Γενικών Διευθύνσεων. Και θα θέλαμε να ζητήσουμε από την εκπρόσωπο της Γενικής Διευθύνσης Δικαιοσύνης, την κυρία Στόλα να παραμείνει μέσα στην αίθουσα προκειμένου να συζητήσουμε το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το οποίο αφορά την ασπίδα προστασία, όπω ονομάζεται, τη ιδιωτική ζωή Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το σημείο λοιπόν ε, θα συζητηθεί και κλεισμένο το θυρών. Οπότε όσοι δεν δικαιούνται να παραμένουν στην αίθουσα, τους ε, παρακαλώ να αποχωρήσουν. Και όσοι βέβαια δικαιούνται να παραμείνουν.